Από τη συζήτηση αυτή συνάγω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο Ιράκ πολύ στενά και ε, να συνοδεύσουμε τη χώρα από την σταθεροποίηση στην ανασυγκρότηση, στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευημερία. Επίσης θα πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία στις διμερείς και πολυμερείς μας επαφές για να ε, διατρανώσουμε και πάλι πόσο επίγον είναι να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και στις ανάγκες του Ιρακινού λαού ε, και στην ε, γενικότερη κατάσταση. Τους επόμενους μήνες έχουμε τις πρώτες ε, διαπραγματεύσεις από την Συμφωνία Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιράκ από τότε που τέθηκε σε ισχύ. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και τη διατήρηση του θέματος αυτού τόσο ψηλά στο θεματολόγιο και στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστούμε Υπουργέ του Πουράινεν, Κίτος. Ε, τώρα κυρίζω τη λήξη τη ε, συζήτηση για το θέμα αυτό. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Πολιτική δήλωση υψηλού επίπεδου των ΕΕ με θέμα την καθολική υγειονομική κάλυψη. Και πριν ξεκινήσει η συζήτηση, να σα ενημερώσω ότι αν θέλετε να ζητήσετε το λόγο βάσει τη διαδικασία ε, και με τη γαλλική κάρτα, να κοιτάξετε να εγγραφείτε κανονικά, ιδάλω με το σύστημα που επιτρέπει στου βουλευτέ να εγγραφούν ηλεκτρονικώ. Και γι' αυτό καλό θα είναι πάντα να, έχει μαζί, να έχετε μαζί σα την κάρτα ψηφοφορία. Εάν θέλετε λοιπόν να εγγραφείτε στην ε, διαδικασία καθιστιά, κάντε το από τώρα, χωρί να περιμένετε το τέλο τη συζήτηση. Ε, για να ξεκινήσουμε, ο λόγος στην Υπουργό του Συμβουλίου, την κυρία Τοπουράιναν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σας ε, επισημάνω ότι το να μιλούμε για την υγεία σε τόσο προχωρημένη ώρα είναι κάπως αντιφατικό. Ε, είμαι στην Ολομέλεια από τις 9 το πρωί και κανονικά αν σκεφτόμασταν την υγεία μας θα έπρεπε τόσο αργά που είναι να αναπαυόμασταν. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να σας μιλήσω και να συζητήσουμε την πρόσφατη ε, διαδήλωση, ε, δήλωση υψηλού επίπεδου που έγινε στις 23 Οκτωβρίου για την καθολική υγειονομική κάλυψη και την προσπάθεια από κοινού να δημιουργήσουμε έναν υγιή κόσμο. Ε, έδωσαν εκεί το παρόν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ηθήνοντες πολιτικής και πρωτοπόροι σε θέματα υγείας. Η υγειονομική, καθολική, καθολική υγειονομική κάλυψη σημαίνει όλοι, ακόμη και οι πιο ευάλωτοι και κυρίως οι πιο ευάλωτοι, να έχουν πρόσβαση στην υγεία όποτε και όπου το χρειάζονται, χωρίς να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες ε, που σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τις ε, υποσχέσεις μας ε, και να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε τέτοιες ε, υπηρεσίες υγείας, ε, βαίνοντα προς μια καθολική υγειονομική κάλυψη και επίσης ε, εξασφαλίζοντας ειδικευμένο προσωπικό υγείας και πρόσβαση σε φάρμακα και εμβόλια σε προσιτές τιμές καθώς και ποιοτικέ υγειονομικές υπηρεσίες. Επίσης, όλες αυτές οι δράσεις πήραν τη μορφή μιας πολιτικής διακήρυξης για την καθολική υγειονομική κάλυψη με την εκπροσώπηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και μάλιστα αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία πριν το 2023 που είναι η διάμεση φάση για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ε, που έχουν ως καταληκτική προθεσμία το 2030. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε λοιπόν τη μεγαλύτερη πολιτική υποστήριξη ώστε το θέμα της υγείας ε, να ε, στοχεύσει προς την καθολική υγειονομική κάλυψη. Έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για υγιή ζωή και διαβίωση ε, προκειμένου οι εθνικές κυβερνήσεις να τηρήσουν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες υγείας των πολιτών τους. Βέβαια το μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει ακόμη για τη σημαντική χρηματοδότηση που απαιτείται από τώρα μέχρι το 2030 για να υλοποιήσουμε τις φιλόδοξες δεσμεύσεις μας. Η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να εξασφαλιστεί μέσω ενός μείγματος ε, ε, εθνικών πόρων και ε, διεθνών μηχανισμών χρηματοδότησης. Αυτό σίγουρα θα είναι το βασικό μας έργο στο μέλλον. Μπορεί να είναι μεγάλη πρόκληση, αλλά η εξοπιστία μας θα διακυβευτεί αν αποτύχουμε. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να τονίσω τον ηγετικό ρόλο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να συνεχίσουν να το διαδραματίζουν στα πλαίσια της καθολικής υγειονομικής κάλυψης σε πολυμερή φόρα. Για το θέμα αυτό ε, δεν θα πρέπει να το θεωρούμε ως κάτι δεδομένο και μας είναι ιδιαίτερα προσφυλέ ζήτημα. Και το 2020 θα είναι η λιδία λίθος, γιατί θα έχουμε την 25η επέτειο της διάσκεψης του Καΐρου του 1994 και της πλατφόρμας του Πεκίνου του 1995 για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να ε, είμαστε πρωτοπόροι ώστε να συνεχίσουμε αμύωτη την πρόοδο που έχει ξεκινήσει πριν από 25 χρόνια και επουδενή ε, να μην επιτρέψουμε μια παλινδρόμηση. Και μάλιστα η ηγετική θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε και στο, στην εκδήλωση υψηλού επίπεδου για, το καθολικό, για την καθολική υγειονομική κάλυψη. Και πραγματικά ε, χαιρετίζω την ε, προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των ε, σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων θα είναι σημαντικό ε, στοιχείο εν ώψη της υλοποίησης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του 2030 και θα πρέπει η άσκηση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων να, είναι προσιτή σε όλους, ώστε η καθολική υγειονομική κάλυψη να γίνει πραγματικότητα μέχρι το 2030, χωρίς αποκλεισμού και χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Φιλανδική Προεδρία δεν θα αφιστεί προσπαθειών για να προωθεί την καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για όλους τους ανθρώπους και κυρίω για του πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας. Και μάλιστα όπου και χρειάζονται και με βάση την προσέγγιση της ευημερίας και της πρόνοιας που ε, υιοθετεί και στερνίζεται και η Φιλανδική Προεδρία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Κίτος. Και τώρα, εξ ονόματο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπο Μίμητσα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε, και κύριοι. Στι 23 Σεπτεμβρίου, η Αρχική Κρατών και Κυβερνήσεων, καθώς και οι Υπουργοί Υγεία, συνήλθαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για πρώτη φορά στα χρονικά για μια συνάντηση υψηλή επίπεδου για την καθολική υγειονομική κάλυψη. Ήταν ένα ερώσιμο η πολιτική τους δήλωση με νέα τόλμη για να δημιουργήσουμε έναν υγιέστερο κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει αυτό το ιστορικό γεγονός τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ αναγνωρίζουν τώρα ότι η υγειονομική καθολική κάλυψη πρέπει να ισχύει για όλους. Η πρόσβαση σε πρόληψη, ε, θεραπεία, αποκατάσταση καθώς και αποθεράπευση και τις σχετικές υπηρεσίες παρηγορητική αγωγή, καθώς και τα ανάλογα φάρμακα. Τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να επενδύσουν σε πρωτογενή υγειονομική κάλυψη, προκειμένου να υπάρχει ε, προσβάσιμη κάλυψη υγείας για γυναίκες και παιδιά, και να ενισχύσουν όσου εργάζονται στον τομέα τη υγεία, ενισχύοντα τι ε, δυνατότητε υγειονομική κάλυψη των διάφορων κυβερνήσεων. Δυστυχώ, βεβαίω, υπήρχε και διχασμό μεταξύ των 100 μελών ε, για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματά τη. Οι κάτω χώρε ε, εξέφρασαν δήλωση εκ μέρου 34 χωρών, υποστηρίζοντα στεναρά την καθολική υγειονομική κάλυψη και για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα που εκπορεύονται από αυτή. Ο ΙΕ μαζί με χώρε, ή είπα μάλλον μαζί με 19 άλλε χώρε διαχώρισαν τη θέση του σε σχέση με τη δήλωση αυτή για μια δυνατότητα ε, αποχώρηση από την ε, σύμβαση στα δικαιώματα αυτά. Η Επιτροπή, μιλώντας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναπιβεβαίωσε την ε, δέσμευσή της, τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την προστασία, καθώς και την πρόθεση όλων των δικαιωμάτων, όλων των πολιτών, για να έχουν το στο δυνατό επίπεδο ε, σωματικής και ψυχολογικής υγείας τα δικαιώματα αυτά είναι σημαντικά για να έχουμε σταθερές και ευμερούσες κοινωνίες, ε, οικονομική ε, ευμάρεια και ασφάλεια. Το να αντιμετωπίσουμε την υγεία ως ένα φαινόμενο καθολικό μαζί με μια ε, προσέγγιση σφαιρική που έχει χρησιμοποιηθεί και στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων θα πρέπει να έχουμε τον παράγοντα υγεία σε όλε τι πολιτικέ τη Ένωση και περνώντα τα σύνορα του απλού υγειονομικού κλάδου. Ε, θα πρέπει να εργαστούμε όλοι ταυτόχρονα για την ισότητα των φύλων, για την σωστή υγειονομική κάλυψη, τον επισκεπτισμό και την επιστηστική ασφάλεια, την αξιοπρεπή εργασία, την προστασία, των περιβάλλων και την ασφάλεια. Αυτά όλα, εάν προωθηθούν, θα μα φέρουν ίσω καλύτερα αποτελέσματα. Υπ' αυτήν την έννοια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει δεσμευμένη για την προώθηση, την προστασία και την εκπλήρωση όλων των προποθέσεων που απαιτούνται για τα δικαιώματα, όλα τα δικαιώματα μαζί με τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά και να συνεχίσει την, την διαρκή εφαρμογή της πλατφόρμας του Πεκίνου, πλατφόρμα δράση που συμφωνήθηκε με τη νέα συνένεση για την ανάπτυξη. Στη σύνοδο του Ναϊρόμπι τον ε, Νοέμβριο θα γιορτάσουμε και θα επαναλάβουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο του, της Διεθνούς Συνόδου για τον Παγκόσμιο Πληθυσμό που είχαν εγκριθεί πριν από 25 χρόνια. Η αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου θα πάρει μέρος σε αυτή τη σύνοδο υψηλού επίπεδου. Η δράση οι δράσει τη Ένωση έχουν δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μεταξύ του 2013 και του 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισέφερε σε περνό από 19 εκατομμύρια ε, που τι έφεραν ει πέρα ε, ε, ε, προσωπικό με Ε, Δεξιότητες. 13 εκατομμύρια βρέφη γεννήθηκαν ε, με... εμβολιάστηκαν εγκαίρως. 600 ε, εκατομμύρια ε, εμβόλια οι μοιράστηκαν για την προστασία από την ελονοσία. Υποστηρίχθηκαμε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Και συνυπογράψαμε μία κοινή δήλωση 200 εκατομμυρίων, ε, ενό προγράμματο εταιρική σχέση 200 εκατομμυρίων ευρώ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία για την παγκόσμια υγειονομική κάλυψη. Ω ε, διεθνή πρωταγωνιστή, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τι χώρε εταίρου στι προσπάθειέ του να χτίσουν ισχυρέ, καλή ποιότητα και ανθεκτικέ υγειονομικέ υπηρεσίε με ε, κατάλληλη πρόσβαση σε όλε τι ιατρικέ υπηρεσίε και την ιατρική κάλυψη. Υπ' αυτήν την έννοια θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε το φιλόδοξο στόχο μας της καθολικής υγειονομικής κάλυψης για όλους ως το 2030. Σας ευχαριστώ. Χβάλα. Κύριε Επίτροπε, αρχίζει ο γύρος των ομιλητών εξ ονόματος των πολιτικών του ομάδων. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η κυρία Μονσεράτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε προχωρήσει πολύ στην καταπολέμηση των βασικών αιτίων θανάτου και νόσων στον κόσμο. Έχει ε, αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο το προσδόκιμο ζωής, έχει μειωθεί ε, η θνησιμότητα των ε, βρεφών και των γυναικών, έχει μειωθεί το AIDS και η ελονοσία. Ωστόσο η πρόοδος στον κόσμο δεν είναι η ίδια 31 χρόνια μεσολαβούν ε, από ε, το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής στο υψηλότερο. 400 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό πόσιμο. Ε, κάθε λίγα δευτερόλεπτα πεθαίνει κάποιος ηλικίας 30-70 ετών από αίτια και νόσους που δεν είναι θανατηφόρες. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι ε, η καθολική υγειονομική κάλυψη μας δίνει μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, αλλά είναι και κινητήρας για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική. Η Ευρώπη είναι παράδειγμα επιτυχίας, όπου έχουμε το καλύτερο σύστημα δημόσιας υγείας. Ε, από την πρωτοβάθμια φροντίδα επενδύουμε. Ε, κάνουμε έρευνα για τις θεραπείες, τις πιο προηγμένες. Έχουμε τους καλύτερους υγειονομικούς ε, και έχουμε ποιότητα και καθολικότητα ε, στην ε, φροντίδα υγείας και στην πρόσβαση θεραπείας. Αυτό που θέλουμε είναι ο τρίτος στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης να γίνει πραγματικότητα παγκοσμίω στην Ευρώπη. Έχουμε δύο σπουδαία εργαλεία και είναι η δύναμή μας για να φτάσουμε στους στόχους μας. Το πρώτο είναι το ευρωπαϊκό μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης και το δεύτερο είναι το μοντέλο διεθνούς συνεργασίας. Ζητώ λοιπόν από τη Φιλανδική Προεδρία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προαγάγει τη συνεργασία μας με άλλες χώρες για να μοιραστούμε τη γνώση, την έρευνα και την πρόσβαση στις θεραπείες. Στην Ευρώπη είμαστε ηγέτες στη διεθνή συνεργασία. Πάνω από 72 δις ε, αφιερώνουμε το χρόνο και πολλά για την υγεία σε προγράμματα. Όπως είναι η πρόληψη και προγωγή της υγείας που αρχίζει από τη διατροφή και μάλιστα από την πρωτοβάθμια φροντίδα και τα αναπτυξιακά προγράμματα συνεργασίας θα πρέπει να κατευθύνονται κυρίως στη μείωση ε, της θρησιμότητας των ε, ε, γυναικών και των βρεφών και επίσης να σταματήσουν οι επιδημίες μεταδοτικές νόσοι και οι θάνατοι να μειωθούν από νοσήματα που δεν είναι θανατηφόρα. Άρα το 2030 θα πρέπει να υπάρχει καθολική υγειονομική κάλυψη σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε συνάδελφοι. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα με το χρονόμετρο που δεν λειτουργεί. Τέλο πάντων, ήταν δικό μα το πρόβλημα, δεν φταίτε εσεί. Καταλαβαίνω ότι ήταν δύσκολο να τηρήσετε το χρόνο της παρέμβασής σας. Το λέω και στο συνάδελφο, για τον συνάδελφο Φεραίρα που είχε ζητήσει γαλάζια κάρτα. Είχαμε ορίσει ότι στον πρώτο γύρο παρεμβάσεων εξ των πολιτικών ομάδων μεταξύ των αντιπροέδρων είχαμε αποφασίσει να μην ε, δίνουμε το δικαίωμα για ερώτηση με γαλάζια κάρτα. Και τώρα ο λόγος του εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκράτων ε, τον, τον, κύριο Φριτσόν, για να λεπτό, κυρία Φριτσόν για 1,5 λεπτό. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Εμεί στην ομάδα των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών χαιρόμαστε για την πολιτική διακήρυξη ψηλού επίπεδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γιατί? Γιατί θέλουμε να υλοποιήσουμε του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε καθολική υγειονομική κάλυψη. Είναι σημαντικό αυτό για να βελτιώσουμε την υγεία των ε, ανθρώπων όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο. Και η πρόσβαση στι υγειονομικέ υπηρεσίε είναι θεμελιώδη δικαίωμα. Όλοι ε, οι συνάνθρωποι μας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικέ υγειονομικές υπηρεσίες ε, όπου και αν βρίσκονται, όποτε τις χρειάζονται, ασχέτως του φίλου τους, της ηλικία τους ή της κοινωνικής τους τάξης. Κανένας δεν θα πρέπει να αποκλείεται από την καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Βλέπουμε όμως δυστυχώς ότι σε πολλές περιοχές του κόσμου δεν έχουν όλοι οι συνάνθρωποι μας πρόσβαση σε ποιοτικές υγειονομικές υπηρεσίες. Δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε πρόσβαση σε υπηρεσίες που αφορούν τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους δικαιώματα. Σε πολλές χώρες του κόσμου οι γυναίκες στερούνται τέτοια δικαιώματα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επομιστούν τις βαρύτατες ευθύνες που έχουν. Θα πρέπει όλες οι γυναίκες να έχουν δικαίωμα στην άβλωση. Το δικαίωμα στην άβλωση είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να αποφασίζει για το σώμα του και εμεί οι σοσιαλιστές θα δώσουμε μάχη ώστε όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες να έχουν ίσα δικαιώματα και όλοι να έχουν δικαιώματα σε ποιοτικέ και ασφαλείς υγειονομικές υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ εκ μέρου τώρα της ομάδας Renew Europe. Το λόγο έχει η κυρία Τριγέ Λενουάρ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική διακήρυξη τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Καθολική Υγειονομική Κάλυψη αναγνωρίζει το σημαντικό αντίκτυπο που έχουν οι περιβαλλοντικέ ε, συνθήκε στην ανθρώπινη υγεία. Η ατμοσφαιρική ρήπαση οφείλεται για 400.000 πρόωρου θανάτου το χρόνο στην Ευρώπη και για πολλού καρκίνου. Επίση, η ρήπαση του νερού και των τροφίμων από τοξικού παράγοντε μπορεί να δημιουργήσει αναπαραγωγικά προβλήματα. Η υπερθέρμανση του πλανήτη διευκολύνει την εξάπλωση των ασθενειών ε, και ε, με τις, μέσω της μόλις από κουνούπια. Και μάλιστα ε, δύο κρούσματα αυτόχθονου ιού Ζήκα βρήκαμε στη Γαλλία. Η καταπολέμηση λοιπόν της κλιματικής απορρίθμισης είναι βασικός άξονας της εξασφάλισης καθολικής υγειονομικής κάλυψης. Έχουμε επίγνωση αυτής της πραγματικότητας και του ηγετικού ρόλου που οφείλει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία απόλυτη και ύψιστη προτεραιότητα. Η Συμφωνία των Παρισίων μάλιστα μας υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στην υγεία είναι από τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Ο πρωταρχικός στόχος της νέας Πράσινης Συμφωνίας θα πρέπει να είναι η ανθρώπινη υγεία και κυρίως η υγεία παγκοσμίω, που θα δημιουργήσει ένα ενάρετο κύκλο μεταξύ τη ανθρώπινη υγεία, ε, τη υγεία του περιβάλλοντο και τη υγεία των ζώων. Στην καταπολέμηση τη υπερθέρμανση του πλανήτη και το μετριασμό τη κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη σωστή διαπαιδαγώγηση των πολιτών, ώστε να αποφύγουμε νέε ανισότητε και στον τομέα τη υγεία που πλήττουν κυρίω του πιο ευάλωτου συμπολίτε μα. Επίση, είναι άρρηκτο ο δεσμό μεταξύ του περιβάλλοντο και τη υγεία. Και αυτό ο άρρηκτο δεσμό θα πρέπει να μα οδηγεί σε σωστή αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πολιτικών με τη χρήση κριτηρίων προσδόκιμου ζωή σε καλή υγεία. Αυτό θα είναι ο καλύτερος δείκτης αποτελεσματικότητα τη νέα πράσινη συμφωνία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία μου, και τώρα εκ μέρου των Πρασίνων Ντεσούτερ για 1,5 λεπτό. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, Uh, Καλωσορίζω ε, την ομιλία του Επιτρόπου Ανδρουκάητης ε, στη συνάντηση υψηλού επίπεδου για την καθολική υγειονομική κάλυψη. Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να αγωνίζεται να γίνει αυτό πραγματικότητα και μέσα στην Ευρώπη. Και χαίρομαι που τόνισε την ανάγκη να ενταχθεί η υγεία σε όλους τους τομείς πολιτικής. Επίσης τόνισε ε, και την προσέγγιση βάσει δικαιωμάτων. Όλα αυτά τα λόγια και οι δεσμεύσει θα πρέπει να γίνουν έργα. Και αυτό γίνεται μόνο με ε, επένδυση στα δικαιώματα στην υγεία για όλους και ίση πρόσβαση. Μόνο έτσι θα υπάρξει καθολική υγειονομική κάλυψη για να είναι πραγματικά παγκόσμια. Θέλω να αφαιρθώ σε κάτι συγκεκριμένο. ω πρόεδρο. Ε, ε, του Φόρουμ για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα ανησυχώ, γιατί κάποιε κυβερνήσει και μεταξύ αυτών και ευρωπαϊκέ αντιτίθεται στα δικαιώματα αυτά και στην ισότητα φύλου ε, και στο αντίστοιχο έγγραφο υψηλού επίπεδου. Ευτυχώ που υπήρχαν και προοδευτικά κράτη και επέμειναν για να μπουν αυτά στην τελική διακήρυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να είναι ενωμένη για να υπερασπίζεται τα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω. Είναι σαφέ ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καθολική υγειονομική χάλυψη χωρί καθολική πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγεία. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μίμητσα και την κυρία Τουπουράινεν για την δική τους ε, στράτευση ε, την υπόθεση αυτή. Ευχαριστούμε, Ντάγκ, συνάδελφε. Και τώρα εκ μέρους της ομάδας ID, η κυρία Παλτασάρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το να εξασφαλίσουμε σε όλου του πολίτε του κόσμου τη δυνατότητα να έχουν υγειονομική περίθαλψη ποιότητα και κατάλληλη αγωγή ασχέτω από την ε, προέλευσή τους και την εθνικότητά του είναι θέμα θεμελιδών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει υγειονομική καθολική κάλυψη. Ωστόσο, σήμερα πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει δικαίωμα για βασικές υγειονομικές υπηρεσίες και κάθε χρόνο πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι ε, κάτω από το όριο της βασικής φτώχειας δεν έχουν πρόσβαση στην ε, βασική ιατρική κάλυψη. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια κατάλληλη νοοτροπία πρόληψης. Τρία σημεία για να πετύχουμε με τους στόχους μας. Πρώτον, να έχουμε τις κατάλληλες πόρους για τις εθνικές ε, υποδομές. Χωρίς ε, υποδομές screening δεν μπορούν να εντοπιστούν εγκαίρως καταστροφικές ε, ασθένειες και επιδημίες. Στην Ευρώπη θα πρέπει να στηρίξουμε όσους ασχολούνται με την πρόληψη και την έρευνα και στις φοχότερες χώρες θα πρέπει να κοιτάξουμε κοινωνικονομικές δονημές για να επιτρέψουμε μια αξιοπαπή ζωή. Έχοντας επίγνωση ότι εκπροσωπούμε την Ιταλία μας που θέλει να έχει μια καθολική ιατρική κάλυψη. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την Ιταλική ε, ιατρική κάλυψη που μπορεί ακόμα να βελτιωθεί. Υπάρχουν πολλές αρχές και χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να τα ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ να σέβεστε το όριο του χρονομιλίας σας. Και τώρα, εκ μέρους της ΓΚΟ, ο κύριος Θερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πάνω από το μισό του πληθυσμού του κόσμου δεν έχει καθολική κάλυψη και βασική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Ε, ο ΙΕ πρότεινε την καθολική υγειονομική κάλυψη εδώ και 10 χρόνια. Όμως αν συνεχίσουμε ως σήμερα δύσκολα θα πετύχουμε το στόχο μας. Η ε, καθολική υγειονομική κάλυψη σημαίνει ότι όλοι και όλες οι κοινότητες θα έχουν τις υπηρεσίες υγείας που τους αξίζουν. Πρόληψη, αγωγή, αποκατάσταση και παρηγορητική αγωγή. και χωρίς οικονομικές δυσχέρειες. Όμω το δικαίωμα στην υγεία είναι θεμελιώδε και οικουμενικό δικαίωμα. Όπω ε, βλέπουμε όμω στην πράξη, δεν θα μπορέσουμε με την εμπορία των υπηρεσιών υγεία, την εμπορευματοποίησή του μάλλον, να πετύχουμε του στόχου μα. Βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σε πολλέ χώρε. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι αποσταχωρήσει που έγιναν, ε, τι αποσταδρομήσει εξαιτία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί το δικαίωμα στην υγεία να είναι θέμα εμπορικό. Θα πρέπει να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα στον χώρο τη συνεργασία για την ανάπτυξη. Πρέπει να κοιτάξουμε το πρόβλημα κατάματα και να δράσουμε. Ε, πρέπει να κάνουμε ακόμη πολλά και γι' αυτό λυπούμαστε που οι βασικέ πολιτικέ ομάδε αυτού του Κοινοβουλίου έχουν απορρίψει την συμμετοχή, με τη συμμετοχή του σε αυτή τη συζήτηση ένα ψήφισμα με συστάσει που θα έπρεπε να εγκρίνει το Κοινοβούλιο αντί για αυτό που έχουμε μπροστά μα. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Χίλια ευχαριστώ. Και τώρα Φράνσεν για 1,5 λεπτό. Η κυρία Φράνσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλά κάνουμε και συζητούμε σήμερα την καθολική υγειονομική κάλυψη και μάλιστα παγκοσμίω είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν καμία πρόσβαση στην υγεία. Αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα παραμένουν πολλοί άνθρωποι που για λόγους οικονομικούς δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία. Παρ' όλα αυτά που έχουν δικαίωμα και ανάγκη, η πολιτική διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών πραγματικά τονίζει ε, έναν ε, στόχο βιώσιμης ανάπτυξης. Κοιτάξτε, υπάρχει το θέμα το περιβάλλοντος. Δεν μπορούμε να συζητούμε για υγεία εάν δεν έχουμε υγιεινό περιβάλλον και προστασία από τοξικές και βλαβερές ουσίες. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι διεθνώς ε, δεν προστατεύονται από τοξικές ουσίες. Όταν είσαι φτωχός ε, αρρωσταίνεις και όταν είσαι άρρωστος γίνεσαι φτωχό. Όπου φτωχό και η μοίρα του, όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Ε, έχουμε τεράστια ευθύνη, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς, για τα θέματα του εμβολιασμού. Το να μην εμβολιάζει σημαίνει κίνδυνο για όλο τον πληθυσμό. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε Ε, να καλύψουμε το κόστος. 600 δισεκατομμύρια χρειάζονται στην Ευρώπη, άρα θα πρέπει να αλλάξουμε ταχύτητα και όχι μία ταχύτητα, δύο να αυξήσουμε. Και επίση το θέμα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας το τονίζω. Συνάδελφοι, ε, είναι μεγάλες οι φιλοδοξίες για το 2030 για να φτάσουμε στους στόχους μας ε, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια και τον απαραίτητο έλεγχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Σέρντας για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρωτοβάθμια, φροντίδα, η υγεία είναι ο πιο αποτελεσματικό τρόπο για να ελοπίσουμε κάποια στιγμή την καθολική υγειονομική κάλυψη. Για να ελοπίσουμε όμω το στόχου βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι το 2030, θα πρέπει να επιταχύνουμε το ρυθμό μας. Και όταν βλέπουμε τη συγκέντρωση των ανθρώπινων πόρων στη Ρηγία, βλέπουμε ότι επικεντρώνονται στις μεγάλες αστικές περιοχές, ενώ οι πιο απομακρυσμένε αγροτικέ αγροτικές περιοχές, όπως οι Αζόρες και το Πόρτο Σάντο, που απέχουν από το κέντρο, είναι εξόχως απόκεντρη περιοχή, ε, το 64% των ε, ε, κατοίκων ε, έχουν μόνο ε, οικογενειακό γιατρό. Το 1 τρίτο των κατοίκων ε, δεν έχουν πρόσβαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να χαράξουν και να εφαρμόσουν πολιτικέ που θα προωθούν την υγεία με περισσότερε επενδύσει στην υγεία και με κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη στις ποιοτικέ υπηρεσίε υγείας. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα κίνητρα ώστε να κρατήσουμε υγειονομικό προσωπικό στι πιο απομακρυσμένε περιοχέ και να εξασφαλίσουμε ε, πρόσβαση και στι εξόχω απόκεντρες περιοχέ σε ποιοτικέ υγειονομικές υπηρεσίε. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Αν δεν επενδύσουμε όμω την υγεία, ε, δεν θα επενδύσουμε ουσιαστικά στην ίδια μα την κοινωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ερώτηση με μπλε κάρτα εκ μέρους του κυρίου Σόκολ. Τη δέχεστε, κυρία Σέρδας. Κύριε Σόκολ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Κυρία Σέρδας, χαίρομαι που αναφερθήκατε σε ένα πρόβλημα που υπήρχε, που υπήρχε από την αρχή, την διαφορά και την ανισότητα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Μακάρι να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική συνοχή. Θα, μπορούσατε, ε, πιστε, θα μπορούσε, πιστεύετε, η πολιτική συνοχή να βοηθήσει ε, τις περιοχές της Ευρώπης που δεν έχουν παρκή πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη όπως είναι οι Αζόρες ή άλλες απομακρυσμένες περιοχές για να βελτιώσουν αυτή την πρόσβαση. Ευχαριστώ. La declaración de la ONU es un gran paso adelante. Miren, en 1986. Παίρνει το λόγο ο κύριο Κασάρε. Έχουμε σημειώσει με μεγάλη πρόοδο. Συγγνώμη, προηγείται η κυρία Σέρντα. Άκουσε ερώτηση με, με την μπλε κάρτα και θα έχει το χρόνο για να απαντήσει. Εγώ είχα το λόγο όμως, λέει ο κύριος Κασάρης. Όχι, συγγνώμη. Εσείς είστε μετά. Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Σέρδας που πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση της μπλε κάρτας του κυρίου Σόκολ. Είστε στον κατάλογο των ομιλητών, αλλά αργότερα, μετά την απάντηση που θα δώσει η κυρία Σέρδας. Ευχαριστώ κύριε Σόκολ για την ερώτηση. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη και να ε, καλύψουν τα κενά τους στην υγειονομική παροχή, στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών. Και Ίσως η πολιτική συνοχή θα βοηθήσει τους πολίτες να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε σωστή και ακόμη πρωτοβάθμια φροντίδα Χρειαζόμαστε ανθρώπινους πόρους, γιατί αν δεν έχουμε ε, γιατρούς, υγειονομικό προσωπικό σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, έτσι στερούμε και από τους πολίτες των απομακρυσμένων περιοχών τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικέ υγειονομικέ υπηρεσίε. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα κυρία Τσε για ένα λεπτό. Λουίς, ευχαριστώ. Η υγεία είναι θεμελιώδης δικαίωμα, όλοι συμφωνούμε. Πώ μπορούμε όμω να βεβαιωθούμε ότι ο κόσμο μπορεί να εξασκεί αυτό το θεμελιώδε δικαίωμα. Σήμερα έχουμε ανάγκε που δεν καλύπτονται και έχουμε και τέτοια παραδείγματα από πολλέ ε, χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ω γιατρό του τομέα τη υγεία, μπορώ να σα πω ότι στην χώρα μου, την Ουγγαρία, η πρόσβαση στην υγεία είναι προνόμιο, όχι βασικό δικαίωμα. Ε, το προσδόκιμο ζωή είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολύ μεγάλε ανισότητε ε, ω προ τον τομέα τη υγεία, ανάλογα με το εισόδημα και την κοινωνική προέλευση. Η πρόσβαση στην υγεία έχει να κάνει μόνο με το δυνατότητα κάποιου να πληρώνει και όχι με τις ανάγκες που έχει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν ότι το σύστημα υγείας είναι τελείως συμπερασματοποιημένο. Ας είμαστε βέβαιοι ότι οι ιατροί και οι νοσοκόμες μπορούν να ε, λάβουν την αξία που του αναλογεί και να είναι ένας πραγματικός πλέον της κοινωνίας μας. Μιλάμε για ένα στοιχείο κοινωνικής προστασία ε, προς την υγεία και θα πρέπει να το ε, καλύψουν όλα τα κατημέλη. Πρέπει η πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προάγει και την υγεία των πολιτών μας. Πρέπει να πιέσουμε τις κυβερνήσεις ώστε να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι πολίτε μπορούν να ασκούν το βασικό του αυτό δικαίωμα, το θεμελιώδε δικαίωμα πρόσβαση στην υγεία, ασχέτω ηλικία, κοινωνική προέλευση, κοινωνικού στάτου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Και τώρα λόγο στην κυρία Κονεσνά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, κάποιοι από εσά θα θυμούνται ότι το 2017 ήμουν ένα από τα πρόσωπα της εκστρατεία για την πρόθωση της υγειονομική καθολικής κάλυψης όλων των πολιτών μέχρι το 2030, που το πρότεινε το Φόρουμ των Ασθενών της Ευρώπης. Τότε καλούσαμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα όλων των ασθενών ασχέτως του που βρίσκονται σε ποιο κράτος μέλος και που κατοικούν Θέλαμε να έχουν υψηλού, ε, υψηλής ποιότητας κάλυψη και πρόσβαση στο σύστημα υγείας, ώστε οι γιατροί, οι ιατροτεχνικές συσκευέ και οποιαδήποτε είδους υπηρεσία χρειάζεται να ήταν κάτι στο οποίο θα, έπρεπε, θα έχουν πρόσβαση όλοι, χωρίς να υπάρχει στιγματισμός των ασθενών που να αποκλείονται από το κοινωνικό σύνολο. Ωστόσο, καμιά από αυτές τις υποσχέσεις δεν τηρήθηκαν από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Ωραίο είναι που στη δήλωσή μας συζητάμε ε, ότι οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κατών και κυβερνήσεων δίνουν, ε, ε, χτυπάνε ένα στην πλάτη του άλλου ε, επενετικά, αλλά δεν έχουν καταφέρει αυτό που ζήτησαν το Ευρωκοινοβούλιο. Καλύτερη κάλυψη όλων των ασθενών που θα πρέπει να το εφαρμόσουν τα ευρωπαικα κρατημέλη. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε. Και τώρα ο λόγο στον κύριο Σόκολ για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Γνωρίζουμε και φαίνεται και από τη συζήτηση ότι υπάρχει συνένεση ότι ε, είναι οικουμενικό και αναπαρατηρεί το ανθρώπινο δικαίωμα η καθολική υγειονομική κάλυψη. Δυστυχώ όμω, ε, πολλοί άνθρωποι δεν απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα στην υγειονομική κάλυψη. Και είδαμε και από προηγούμενε συζητήσει ότι υπάρχουν πολλέ διαφορέ, ακόμη και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική κάλυψη υπάρχει διαφορά μεταξύ των αστικών κέντρων του Βορρά σχέση με τις πόλεις του Νότου, ε, ε, τη διαφορά μεταξύ Ανατολής ε, και Δυτικής, Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης ή διαφορά μεταξύ αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε όχι με πολιτική λιτότητα να βελτιώσει την κάλυψη. Δυστυχώ είχαμε δρακόντια μέτρα και μάλιστα μέσω οικονομική κρίση, κάτι που είναι αντιφατικό με το στόχο τη καθολική υγειονομική κάλυψη. Χαίρομαι πάντω που και το ΕΛΚ βρήκε την κατάλληλη στιγμή να θέσει το θέμα της καθολικής υγειονομικής κάλυψης στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε το συντομότερο δυνατό να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Έχουμε πολλούς μηχανισμούς που μπορούν να μας βοηθήσουν να διορθώσουμε αυτές τις ανισότητες στην υγειονομική κάλυψη. Ένας από τους μηχανισμούς αυτούς είναι η πολιτική συνοχή που εδράζεται στην αρχή της αλληλεγγύης ώστε οι λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχές να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να πλησιάσουν τις πιο ανεπτυγμένε περιοχές και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υγειονομική κάλυψη. Με ισχυρή λοιπόν πολιτική συνοχή μπορούμε να φέρουμε την υγεία στις βασικές προτεραιότητες ε, ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε αυτό το πραγματικά οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα τη καθολικής υγειονομική κάλυψης να ε, μπορούν να το απολαύσουν όλοι οι συμπολίτε μα. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριο Τσοχαντάρου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε και κύριοι. Εγώ είμαι γιατρός ε, και εντατικολόγος ε, ε, ήμουν στο Νιου Τζέρσι και πραγματικά ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτά τα πράγματα και η καθολική υγειονομική κάλυψη είναι τεράστιο ζήτημα. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα η πρόσβαση στην υγεία. Είναι όμως και πολλοί οι φραγμοί που πρέπει να ξεπεραστούν. Ε, η αγωγή υγεία. πρέπει να είναι μάθημα στο σχολείο, να γνωρίζει ο καθένα, τι πρέπει να κάνει για να ζει με τρόπο υγιεινό και όχι μόνο για το περιβάλλον. Επίση, υπάρχει και άλλο εμπόδιο οικονομικό που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. σω θα πρέπει να σκεφτούμε μαζί μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σήμα υγεία και να υπάρχει καθολική περίθαλψη παντού στην Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο. Ένα πρόγραμμα υγείας για τις γυναίκες, για παράδειγμα. Για έγκαιρη διάγνωση ε, του καρκίνου. Επίσης, ε, η αναπαραγωγική υγεία θα πρέπει να παρέχει ε, ε, κατά πολέμηση του καρκίνου, ε, δωρεάν εξετάσεις εγγύων κτλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσιχοντόρου και τώρα ο κύριος Αγιορίνο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο ΙΕ ενέκρινε πολιτική δήλωση για την καθολική και νομική περίθαψη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Έτσι ανέλαβε σωματική δέσμευση επισήμως διότι πρέπει να έχουμε απτά αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα και θα πρέπει το δικαίωμα στην υγεία για όλους να είναι κάτι το αναντήρητο. Αλλά δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Το να έχουμε μια πραγματική καθολική υγειονομική κάλυψη σημαίνει ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες ποιότητας, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες. Το ίδιο και για τα φάρμακα και τα εμβόλια που θα είναι δραστικά και αποτελεσματικά. Θα υπάρχει το ίδιο για τους κοινωνικού λειτουργούς, τους γιατρούς και τους νοσοκόμε, τους οποίους όλοι θα εξασφαλίζουμε εξωπρεπή εργασία. Γι' αυτό χρειάζεται μια ριζική αλλαγή πορείας σε πολλές περιπτώσεις και κυρίως σημαντικές επενδύσεις. Επενδύσεις που δεν σημαίνουν κόστος, είναι επένδυση. Αυτή η κοινότοπη η αρχή είναι κάτι που πρέπει να το επιβεβαιώνουμε και με τη στάση μας και με τις επιλογές μας για να εξασφαλίσουμε ε, σωματική και ψυχολογική καλή υγεία για άντρε και γυναίκε. Ευχαριστούμε κύριε Μαγιορίνο. Υπάρχει γαλάζια κάρτα από τον κύριο Σόκολ. Τη δέχεστε κύριε Σόκολ. Ευχαριστώ. Ε, αναφέρατε πολλά πράγματα που πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν για να λυθεί το πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρμόδια για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση και κονδύλια για να ε, επηρεάζει ε, την άσκηση πολιτικής υγείας στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ, Ε, σε σχέση με την ερώτηση, είμαι πεισμένος πω ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει πόρου και επιπλέον θα πρέπει να είναι συνεπής με τον εαυτό της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κοινωνικός πυλώνας ήδη προβλέπει αρχές και συγκεκριμένες επιλογές. Τις έχει ήδη καταδείξει. Το θέμα είναι να μην τα θυμόμαστε όλα αυτά τη στιγμή που απλώς ε, την προσοχή μας τραβάνε οι πιο ευπαθείς ε, και όταν έχουν επιβληθεί σε αυτούς πολιτικές λιτότητας θα πρέπει να αποφασίζουν ε, ε, οι συνθήκες της πραγματικότητας τι πολιτική στα χαράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να συζητάμε με πυγμή και αποφασιστικότητα. Ευχαριστούμε κύριε Μαγιορίνο. Ο κύριος Γκονθάλης Χασάρης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η διακήρυξη του ΟΗΕ είναι ένα βήμα πρόοδου. Το 1987 ο Ερνές Ιούκ στην Ισπανία, ε, καταλανός, ε, ε, εισήγαγε την καθολική υγειονομική κάλυψη. Μετά από 25 χρόνια η κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος τον απέσυρε αυτό το νόμο και έβαλε δυναμή της στα θεμέλια του συστήματος. Εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς κάλυψη με αύξηση των επιδημιολογικών κινδύνων και ε, χιλιάδες νέοι που μετανάστευσαν λόγω κρίσης Έμεινα χωρίς ε, κάλυψη. Το 2018 η κυβέρνηση, η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσε θα αποκατέστησε τον νόμο. Γιατί τα λέει αυτά. Δεν αρκούν μόνο οι διακηρύξει. Θα πρέπει να ε, ε, προσέχουμε και να επαγρυπνούμε τι γίνεται στα δεξιά για να μην επανέλθει η περικοπή τη υγεία στην Ευρώπη. Το δικαίωμα τη προστασία υγεία δεν καταλαβαίνει ούτε από σύνορα, από θρησκεία, από φιλή, από φίλο, από ηλικία και δεν σημασέβεται. Θα πρέπει να επανέλθουμε στην πρόοδο και πάντα να υπερασπιζόμαστε και να προασπίζουμε αυτές τις ιδέες. Ευχαριστώ κύριε Κωσάλης Κασάρες. Ε, γαλάζια κάρτα έχει η κυρία Μονσεράτ, τη δέχεστε. Παρακαλώ. Η Ισπανία ποτέ δεν σταμάτησε να έχει ε, καθολική δωρεάν υγειονομική κάλυψη για όλους τους Ισπανούς. Ψεύδεστε. Ε, Απάντηση. Θέλω να πω στην κυρία Μονσερά που διατέλεσε και Υπουργό Υγείας ότι βγάλατε διάταγμα ε, ναι, αλλά για όλους τους Ισπανούς. Ναι, γιατί μια υπουργό σαν εκείνη προσπάθησε να κάνει διακρίσεις απέναντι σε εκείνους που δεν ήταν Ισπανοί. Οι, ε, Ισπανοί νέοι που είχαν φύγει πάνω από τρεις μήνες έμεναν χωρίς κάλυψη. Ερχόντουσαν νέες ε, να γεννήσουν στη χώρα μας και δεν μπορούσαν γιατί τους είχατε αφαιρέσει το δικαίωμα. Ξέρω ότι δεν το κάνατε εσείς προσωπικά, αλλά είστε συνυπεύθυνοι γι' αυτό. Και μάλιστα σήμερα στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδρίτης αποπειράθηκαν να κάνουν το ίδιο στις πολιτικές ε, υγείας που έχουν μεταφερθεί σε επίπεδο αυτόνομης περιφέρειας οι αρμοδιότητες. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται λοιπόν εδώ η συζήτηση αυτή. Και τώρα να ξεκινήσει η διαδικασία του ΚΑΤΣΤΙΑΕ. Έχω ένα μόνο αίτημα. Η κυρία Ward. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι υπερήφανη που προέρχομαι από, μια πολιτική, από ένα πολιτικό κόμμα που δημιούργησε την Εθνική Υπηρεσία Υγεία. Το Εργατικό Κόμμα κατοχύρωσε το καθολικό δικαίωμα για τους πάντες, από το Λίκνο μέχρι τον Τάφο. και όλοι είχαν δικαίωμα σε δωρεάν υγειονομική κάλυψη και το κάναμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν είχαμε ακόμη τα συσίτια. Όταν ένα κόμμα ε, διαγράφει τα ε, το κόστος της συνταγογράφησης ε, και ε, φέρνει την υγειονομική κάλυψη σε δωρεάν επίπεδο, τότε βάζει τον άνθρωπο μπροστά από τις πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες. Δυστυχώς δεν έχουν όλοι όμως τέτοιο δίκτυο ασφαλείας παντού. Πάντως είμαι περήφανη που η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στήριξε 57 εκατομμύρια γυναίκε να χρησιμοποιήσουν αντισύλληψη, εμβολία σε 13 εκατομμύρια παιδιά και έδωσε 11 ε, εκατομμύρια θεραπείες για τον ιό του AIDS και ε, μοίρασε 600 εκατομμύρια κουνουπιέρες για την πρόληψη της ελονοσίας. Μόνο έτσι θα υλοποιήσουμε σταδιακά την καθολική υγειονομική κάλυψη και θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χίλια ευχαριστώ. Δεν έχω λάβει άλλα για την διαδικασία Κατσιάη, οπότε να κλείσει η συζήτηση και θα ξαναδώσω τον λόγο στον, στον Επίτροπο Μίμητσα. Παρακαλώ, Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίε και κύριοι βουλευτές. Σα ευχαριστώ για τη ζωντανή και πολύ χρήσιμη συζήτησή σα. Νομίζω ότι προέκυψε με σαφήνεια ότι όλοι συμμεριζόμαστε τις αξίες τη καθολικότητα, τη ποιότητα και τη ισότητα για την πρόσβαση στις ε, υπηρεσίες υγεία. Κάτι που είναι και ο απότερο στόχο τη καθολική υγειονομική κάλυψης. Όλα τα συστήματα υγεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να το υιοθετήσουν. Η έγκριση τη δήλωσης του ΟΗΕ είναι ένα σημαντικό εργαλείο καθώ προωθεί βασικέ αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι σημαντικέ δεσμεύσει των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα θα λάβουν σάρκα και ωστά. Θα μεταφραστούν σε πραγματικέ πράξει σε όλο τον πλανήτη. Ε, υπ' αυτήν την έννοια, η δήλωση περιλαμβάνει και έναν επίσημο μηχανισμό αναθεώρηση που θα μα επιτρέψει να ε, σπουγομετρήσουμε την πρόοδο που θα έχει, κατά, ε, θα, έχουμε, θα έχει γίνει μέχρι το 2020 και 2022. Έτσι θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την προσέγγιση μας και τις προσπάθειές μας προτού συναντηθούμε για μια άλλη επίσημη σύνοδο υψηλού επίπεδου το 2023 και να δούμε πώς πήγε η υλοποίηση των υποσχέσεων που είχαν δοθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις χώρες οι οποίε προσπαθούν να επιτελέσουν πρόοδο προ την κατεύθυνση τη καθολική υγειονομική ε, κάλυψη με εξωτερικέ μα δράσει. Μαζί με την εξωτερική διάσταση όλων των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών και τι εταιρικέ μα σχέσει με τρίτε χώρε σε περιφερειακό και διεθνέ επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Και τώρα ο λόγο στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου, την κυρία Τουπουράινεν, για να κλείσει αυτή η μαραθώνια συζήτηση που έβαλε σε δοκιμασία την ίδια μας την αντοχή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χίλια ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη κυρίες και κύριοι. Για να κλείσουμε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πάρα πολύ χρήσιμη συζήτηση και να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία μας, η Φιλανδική Προεδρία, δεν θα αφιστεί προσπαθειών για να εξακολουθεί να προάγει την καθολική υγειονομική περίθαλψη ε, που χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι. Είναι ένα δικαίωμά τους, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων. Και αυτό νίκει στην προσέγγιση της οικονομίας ε, του ΕΦΖΙΝ που έχει εισαγάγει η Φιλανδική Προεδρία με βιώσιμη επένδυση. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ανάγκες και τα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών, μεταξύ αυτών αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία και δικαιώματα. Εμείς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον ΟΗΕ υποστηρίζουμε την πολυμερή προσέγγιση και μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αντίστοιχη διάσκεψη και την πλατφόρμα του ε, Πεκίνου που θα γίνει το 2020. Σας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας και νομίζω ότι έχει ώρα να πούμε ένα καλή νύχτα και κοιμηθείτε καλά γιατί κάνει καλό και στην υγεία σας δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω. Σας ευχαριστώ πολύ και στα φιλανδικά κήτος. Λήξη τη συζήτηση, επόμενη συνεδρίαση θα γίνει αύριο, 5η 24 Οκτωβρίου 2019. Ε, έχει δημοσιευθεί η μερίσια διάταξη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας νύχτα σε όλους συνάδελφοι.